Good morning, ladies and gentlemen. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ήτρε για το 2018, τις καλύτερες ευχές μας για καλή χρονιά σε όλους ε, για αυτή την περίοδο. Να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, Μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Δεν βλέπω κάποιον να έχει σχόλια. Εγώ δεν έχω κάποια ανακοίνωση. Έγκριση ήταν πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων, 6 Νοεμβρίου 2018. Αν δεν υπάρχουν ενστάσεις μέχρι το πέρας της συνεδρίασης, θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται τα πρακτικά. Και πάμε στο σημείο 4. Δημιουργία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας με σκοπό τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της ικανότητας καινοτομίας της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ε, πρόκειται για σχετικά νέο ζήτημα και μάλιστα ξεκίνησε από τους συναδέλφους από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή ΣΕΝΤΕ ε, συνάδελφοι που συζητούσαν ε, το θέμα εδώ και κάποιους μήνες, σχεδόν δύο χρόνια. Και φυσικά το βιομηχανικό σκέλος ε, της ιδέας τους είναι της αρμοδιότητάς μας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν το θέμα αυτό. Η συγγήτρια, η Φρανσουάς Γκροστέτ, θα λάβω ε, το λόγο να πω ότι η σημερινή συζήτηση θα γίνει για να συζητήσουμε τις 472 τροπολογίες ε, που υπέβαλαν τα μέλη στις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, υπάρχουν και φυσικά και τροπολογίες στο σχέδιο έκθεσης. Όπως θα θυμάστε, η κυρία Γκροστέτ ε, παρουσίασε στις 27 Νοεμβρίου την έκθεσή της ε, στη συνεδρίαση της Επιτροπής μας και τώρα θα συζητήσουμε τις τροπολογίες. Να δώσω το λόγο στην κυρία Γκροστέτ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που υπέβαλαν τις τροπολογίες. Όπως υπενθυμίσατε, Έχουμε σημαντικό αριθμό τροπολογιών. Οι συνάδελφοι υπέβαλαν 417 ε, και συνολικά έχουμε 472. Γεγονός που δείχνει ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η βιομηχανική πρωτοβουλία και η συνεισφορά φυσικά της Επιτροπής μας. Υπενθυμίσατε κι εσείς ε, κύριε Πρόεδρε ότι αυτή είναι η αρχή μιας πιο συγκεκριμένης συζήτησης για την άμυνα γιατί θέλουμε να υποστηρίξουμε και τη βιομηχανική προσπάθεια μετά το στάδιο της έρευνας για το 2019 και το 2020 ώστε να έχουμε μια ευρωπαϊκή ε, βιομηχανία άμυνας που θα είναι πιο καινοτόμος και πιο ανταγωνιστική φυσικά. Όπως είπε ο Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Ζαν Κλωτ η Ευρώπη δεν μπορεί και δεν πρέπει να ε, δίνει υπεργολαβία βία την ασφάλεια και την άμυνά τη, Πρέπει λοιπόν να υπάρχει καλύτερη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τα προγράμματα. Ε, να πω αμέσω στου συναδέλφους ότι υπέβαλαν τροπολογίε ότι προφανώς ε, ε, σκοπεύω να λάβω υπόψη όλες αυτέ τι τροπολογίε. Ε, θα πρέπει να εργαστούμε σκληρά και γρήγορα, αλλά με αποτελεσματικά ζητά προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό, διότι μας πιέζουν όπως γνωρίζετε και οι προθεσμίες και πρέπει να τις στηρίσουμε οπωσδήποτε. Να ευχαριστήσω λοιπόν εκ των προτέρων τους συναδέρφους για τη συμμετοχή τους ε, στην όλη αυτή τη δουλειά. Κάποια σημαντικά σημεία τώρα. Όσον αφορά τα ποσά, προβλέπονται 500 εκατομμύρια ευρώ. Κάποιοι μπορεί να πούνε ότι δεν είναι αρκετή, τα κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι είναι υπερβολικά μεγάλο το ποσό. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ λογικό για έργα άμυνα. αποτελούν μια καλή βάση για να ξεκινήσουμε. Βεβαίως υπάρχει και συμμετοχή των κρατών μελών, η οποία θα είναι απαραίτητη. Ε, και είναι απαραίτητο να επιβεβαιώσουμε αυτό το ποσό το οποίο θα επιτρέψει τη χρηματιδότηση αρκετών προγραμμάτων και να υπάρχουν και κίνητρα ε, χάρη σε αυτό για συνεργασία. Θα πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε τουλάχιστον ε, να μην υπάρχουν αλλαγές στον προπολογισμό και να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια από το τον προϋπολογισμό. Πρέπει να υποστηρίξουμε επίσης την ε, ε, βιομηχανική και τεχνολογική βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χρηματοδότηση πρέπει να πάει σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, διότι πρόκειται για κοινοτική χρηματοδότηση. Οι συμπολίτε μας δεν θα αντιληφθούν πώς μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι ευρωπαϊκές με ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτό βέβαια δεν αποτρέπει τη συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις οι οποίες θα είναι εκτό Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια ε, του των ε, ε, έργων του προγράμματος. Ε, και φυσικά δεν απαγορεύει σε καμία περίπτωση στα κράτη-μέλη να συνεχίσουν τη συνεργασία που θεμούν εκτός του προγράμματος. Το πρόγραμμα αυτό δεν έχει στόχο να υποκαταστήσει τα προγράμματα των κρατών μελών. Πρόκειται για κάτι το οποίο είναι εντελώς συμπληρωματικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό βεβαίως να υπάρχουν στρατηγικές εταιρικέ συμπράξεις, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε η Ευρώπη να υποστηρίξει τη βιομηχανία της ώστε να έχουμε μια πραγματική στρατηγική αυτονομία, κάτι το οποίο είναι και το απαραίτητο και αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε. Τέλος, για να δώσουμε κίνητρα για νέες συνεργασίες και κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις ε, διάμεσου μεγέθους επιχειρήσεις, ε, πιστεύω ότι θα πρέπει ε, να κάνουμε τις προσπάθειές μας. Πιστεύω ότι κάθε κράτος μέλος προσπαθεί και νομίζω ότι αυτό αναγνωρίζεται και από το Συμβούλιο. Ε, υπάρχουν κίνητρα λόγω αυτού του κονδυλίου ώστε να προσπαθήσουν τα κράτη-μέλη και πρέπει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, να μπορούν να συμμετέχουν. Ε, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι συνεργάζονται με τις μεγάλες επιχειρήσεις ε, εξοπλισμών ε, σε Καθεστώ υπεργολάβου, αλλά θα πρέπει ο καθένα να έχει δυνατότητα να συμμετέχει. Θα πρέπει λοιπόν ε, να ε, ενισχύσουμε τη διασυνοριακή συνεργασία εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να ε, επιβραβεύσουμε τι επιχειρήσει που επιδεικνύουν καινοτομία και αριστεία. Αυτό είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Για να μπορέσουν να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο κράτη-μέλη, πρέπει τα κριτήρια να είναι ευέλικτα. Τα κριτήρια των τρων απαραίτητων επιχειρήσεων από δύο τουλάχιστον κράτη-μέλα θεωρώ ότι είναι απαραίτητο αν πραγματικά θέλουμε να παρουσιάσουμε νέα προγράμματα. Γνωρίζω βεβαίω ότι θα γίνουν συζητήσει και για τον αριθμό των κρατών μελών, αλλά θα το συζητήσουμε. Θέλω κυρίω να ακούσω και τι έχετε να πείτε. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να βρούμε μια φιλόδοξη συμφωνία για να ξεκινήσουμε πολύ γρήγορα τι διαπραγματεύσει και να φροντίσουμε το πρόγραμμα αυτό να ε, τεθεί σε εφαρμογή από 1η Πρώτου του 2019, όπω το επιθυμεί και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φυσικά ε, με τα χαρά σας συνεργαστώ μαζί σας και κυρίως θα ακούσω τι έχετε να πείτε ε, κειμένου να προσπαθήσουμε να έχουμε και μια σύγκληση απόψε. Ευχαριστώ. Uh, thank you very much, Madam, uh, for your... Ευχαριστούμε πολύ την ε, εισηγήτρια. Ας ξεκινήσουμε τώρα τη συζήτησή μας. οι ισχυώδεις συγητές, ο κύριος Ποχ, δεν είναι εδώ, ο κύριος Μαχτά. Ναι, πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Με την ευκαιρία, καλή χρονιά σε όλους αυτούς που ακόμα δεν είχαν την ευκαιρία να τους ευχηθώ. Εδώ δεν παρουσιάζω βεβαίως την δική μου προσωπική τοποθέτηση, σχετικά με το κατά πόσον πρέπει να υποστηρίξουμε την ε, περαιτέρω επέκταση των οπλικών συστημάτων, αλλά ε, σχετικά με το αν πρέπει να έχουμε στρατηγική αυτονομία ή όχι. Αυτό είναι το βασικό θέμα και επ' αυτού είμαστε αρκετά θετικοί, όπως και να έχουμε τη δυνατότητα ενίσχυσης της καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας ε, στον τομέα αυτό, ο οποίος δοκιμάζεται από τον διεθνή ανταγωνισμό. Βεβαίως, <clears throat> κάποια στοιχεία τα οποία κατά την άποψή μας χρήζουν διευκρίνησης είναι η δικαιούχη η επιλεξιμότητα μάλλον σε αυτά τα προγράμματα. Θα ήθελα να επιμείνω στις ε, συνεργασίες που έχουν οι επιχειρήσεις εκτός Ευρώπης ως προς το θέμα της μεταφοράς τεχνολογίας. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί εκεί μπορεί να έχουμε και καταχρήσεις και λάθη και προσπαθώντας να κερδίσουμε μια πλεονεκτική ανταγωνιστικά θέση πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί απέναντι σε τρίτες χώρες. Δεύτερον, η αιρεσιμότητα των προγραμμάτων αυτών οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον 25 που εδώ συμμετέχουν, πρέπει να είναι συνεπείς. Δηλαδή για τους υποψηφίους χρηματοδότησης ή επιλογής οπλικών στιμάτων, δεν θα πρέπει τελευταία στιγμή να επιλέγουμε άλλον προμηθευτή. Επίσης η πνευματική ιδιοκτησία στα πλαίσια προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται ή στο πλαίσιο αυτό, όλα αυτά είναι υπό την ευθύνη των κρατών μελών, ώστε καθένα να μπορεί να διατηρήσει αυτήν την πλεονεκτική θέση της ανταγωνιστικότητας που μας φαίνεται ουσιοδέστατη. Τώρα, 500 εκατομμύρια είναι πολύ, είναι λίγο. Υπάρχουν διάφορες τοποθετήσεις ο κεντρικός άξονας πάντως και εδώ θα συμφωνούσα με την κυρία Γκοστέτ είναι το σκεπτικό να έχουμε ένα συντονισμό και εν πάση περιπτώσει μια συνεργασία ευρωπαϊκή σε ένα παγκόσμιο διεθνές πλαίσιο που αυτή τη στιγμή είναι κάπως ανισόρροπο. Δεν μπορούμε να αφήνουμε την πρωτοβολία μόνο σε κάποιους. Η βασική λοιπόν ιδέα είναι εδώ να θεωρήσουμε ότι όλοι μπορούν να υποφεληθούν αυτής της καινοτόμου τεχνολογίας προκειμένου να διατηρήσουμε ένα σημαντικό διεθνή ρόλο στα θέματα στρατηγικής και άμυνας. Αυτά είναι τα προκατακτικά μου σχόλια. Έχουμε υποβάλει μαζί με κάποιους συναδέλφους κάποιες τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Τώρα, ε, για το CCR παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, λέει ο κύριος ε, Κρασνοντεύσκη. Να προσθέσω και τις δικές μου ευχές ε, για καλή χρονιά. και ελπίζω να έχετε επανέλθει απολύτως <clears throat> γιατί θυμάμαι ότι είχατε δοκιμαστεί λίγο από κάποια θέματα υγείας παρόλα αυτά είχατε ολοκληρώσει και τις ψηφοφορίες την τελευταία φορά. Τώρα, για τις ε, τροπολογίες ε, και για την έκθεση, ε, εγώ σημειώνω ότι οι τροπολογίες έρχονται από τελείως διαφορετικές πολιτικές ομάδες που αποσκοπούν να βελτιώσουν το κείμενο, να υπογραμμίσουν κάποια θέματα που είναι σημαντικά και θα ήθελα να εκφράσω την συμφωνία μου προς αρκετές από αυτές. Υπάρχει ένα στοιχείο που είναι πάρα πολύ σημαντικό. <clears throat> Πρέπει να οδηγηθούμε σε μια καλή στρατηγική βάση για το αμυντικό τομέα στην Ευρώπη. Αυτή η θέση εκφράζεται. Υπάρχουν και οι τροπολογίες του κυρίου Μπόνι, του κυρίου Κουρουμπάσοφ και άλλων που πηγαίνουν προς την κατεύθυνση αυτής, αυτού του σχολιασμού. Θα πρέπει λοιπόν αυτό το σκεπτικό να εκφράζεται. Επίσης, ε, μιλούμε για κάποιες νέες μορφές συνεργασίας ε, μεταξύ φορέων της βιομηχανίας. Αλλά εδώ μιλούμε για επιχειρήσεις και φορείς που ήδη συνεργάζονται πάρα πολύ καλά μεταξύ τους εδώ και πολλά χρόνια. Εδώ Λίτς, Βέρνερ και άλλοι έχουν υπογραμμίσει αυτό το στοιχείο. Αλλά και αυτή είναι μια πολύ γόνιμη αν θέλετε κατεύθυνση. Τώρα σχετικά με την αύξηση του αριθμού των κρατών μελών που θα ήταν έτοιμα να συνεργαστούν ε, σε, στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων με συγχωρείτε προγραμμάτων. Ίσως να είναι τρία και όχι μόνο δύο τα κράτη-μέλη που έχουμε ήδη. Και εδώ θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τις επιχειρήσεις μέσης κεφαλαιοποίησης και επ' αυτού έχουν υποβληθεί οι τροπολογίες και κάτι ακόμα επί του οποίου θα μπορούσε κανείς να δώσει μεγαλύτερη προσοχή και θα μπορούσαμε να το μελετήσουμε και μεταξύ των σκιωδών είναι το θέμα του ορισμού των οργανισμών που θα έχουν την πιστοποίηση αν θέλετε να συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά. Είχαμε τα θέματα του ορισμού της ευρωαϊκής επιχείρησης, ε, είχαμε τα θέματα της, του συντονισμού και της ομαδοποίησης των ε, επιχειρήσεων που ασχολούνται με τα αμυντικά στην Ευρώπη. Δεν πρέπει να έχουμε διακρίσεις κατά συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Και κάποια άλλα στοιχεία ίσως να οδηγούν κάποια ερωτηματικά, ιδιαίτερα στα θέματα της ε, χρηματοδότησης και της αρμοδιότητος των κρατών μελών Τη κατανομή αρμοδιότητα, δηλαδή μεταξύ κρατών μελών και κομισιών, είμαι βέβαιο ότι θα επαστρέψουμε σε αυτά εν ευθέτω χρόνο. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Η κυρία Βέρινγκ που εκπροσωπεί τον κύριο Ρίκε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και πολύ καλή χρονιά σε όλους. Η Ντομινίκ ο Ντομινίκ δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ το πρωί καθότι προεδρεύει στην Τραν αλλά έχει επανειλημμένος πει ότι υποστηρίζει τη δουλειά αυτή και την χαιρετίζει. Υπάρχει ένα βασικό επιχείρημα, μία βασική θέση που θέλει να εκφράσει ο Ντομινίκ σχετικά με τους στόχους του προγράμματος, ιδιαίτερα έχοντας ε, εξετάσει και τις τροπολογίες. <clears throat> Υπογραμμίζει λοιπόν ότι αυτό το πρόγραμμα αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της ανταγωνιστικότητας των αμυντικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει να συγχέουμε την πρωτοβουλία αυτή με τις πολιτικές διεθνούς συνεργασίας. Ο Ντομινίκ είναι απολύτως υπέρ της ενίσχυσης συνεργασίας με σημαντικούς ευρωπαϊκούς εταίρους όπως το Ηνωμένο Βασιλείο μετά τον Brexit και άλλα μέλη του ΝΑΤΟ αλλά δεν είναι αυτό το σημείο για να εξετάσουμε κάτι τέτοιο. Ο τίτλος του προγράμματος τα λέει όλα από μόνος του. Βιομηχανική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα, χρηματοδότηση για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να θέλουμε αυτό να είναι ένα μέτρο προτεξιονισμού. Εδώ πρέπει να αναπτύξουμε ένα πρόγραμμα που θα κάνει, θα βοηθήσει την Ευρώπη να κινηθεί προς τα εμπρός. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας. Ο κύριος Πουτικόφερ, εξ ονόματος των Πρασίνων τώρα. Happy New Year. Καλή χρονιά. Δεν ήθελα. Ήταν για να σας ξυπνήσω όλους αυτό. Ο θέμα που έχουμε στον τομέα της άμυνας είναι η αποτελεσματικότητα. υπάρχει υπερβολική βιομηχανική παραγωγή, η οποία προστατεύεται εδώ και πάρα πολύ καιρό για εγωιστικούς, περιφερειακούς ή εθνικιστικούς λόγους, η οποία είναι να αντιμετωπίσουμε και τις ε, προκλήσεις αποτελεσματικά. Η περαιτέρω αύξηση των βιομηχανικών ε, δυνατοτήτων στον τομέα είναι λανθασμένος στόχος. Θα πρέπει να τον απορρίψουμε αναφανδών και μάλιστα ε, οι, οι ομάδες πίεσης οι οποίες θα λάβουν ε, τις όλες διαδικασίες που τους μοιράζει χρήμα. Και αυτό από μόνο του είναι διεφθαρμένο ως ιδέα. Η θέση μας είναι να είμαστε περισσότερο φιλόδοξοι να πάμε προς την κατεύθυνση στις 60 περίπου τροπολογίες που υποβάλαμε. Προωθούμε μια εναλλακτική ε, λύση, ένα εναλλακτικό μοντέλο συνεργασίας για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της άμυνας. Ε, δεν είμαστε αντίθετοι στη συνεργασία στον τομέα της άμυνας. Ε, θέλουμε να τον ενισχύσουμε και θέλουμε καλύψουμε όλα τα στενά εθνικά συμφέροντα και να βοηθήσουμε και τον ευρωπαϊκό αμυντικό τομέα ταυτόχρονα. Προτείνουμε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσφέρει τις υπηρεσίες της στα κράτη-μέλη και να βοηθήσει στη διοργάνωση των ε, κοινών αμυντικών προγραμμάτων. Πραγματική μεγάλη επιρροή ε, στην ανάπτυξη του τομέα από τότε που συστήθηκε ε, πριν από περίπου 15 χρόνια πλέον προτείνουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως παράγοντες που οργανώνουν και παρακολουθούν την εσωτερική αγορά να παρακολουθεί την Δυστυχώ μα συγχωρείτε, η ελληνική καμπίνα πρέπει να κλείσει γιατί δεν υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι λόγω ασθενεία. Και... Technology, like cluster munitions, I don't have to list all of that. We imply you to not change the goal, but change the way on which we try to attain the goal of more um, the Council that has already adopted its position. After identifying six criteria, the Council then writes, non-fulfillment of any of these criteria shall not be considered eliminatory. Thank you very much. We don't care for the... Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχηθώ να έχουμε ένα καλό και παραγωγικό νέο έτος. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, κατά την άποψη τη ΓΚΟΕ ε, είναι ξεκάθαρο πως το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδίου για την ε, οικοδόμηση μια στρατιωτική ένωση. Θέσει που υποστηρίζεται δυστυχώς από την εισηγήτρια όσο και από την πλειοψηφία των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί. Η δική μα πολιτική ομάδα η ΚΟΕ τοποθετεί ε, θέσει που υποστηρίζεται δυστυχώ από την εισηγήτρια όσο και από την πλειοψηφία τροπολογιών που έχουν κατατεθεί. Η δική μα πολιτική ομάδα, η ΚΟΕ, τοποθετεί ξεκάθαρα ενάντια σε αυτό το επικίνδυνο εγχείρημα. Στην πρόταση που έχει κατατεθεί, ζητείται να γίνουν επενδύσει στον τομέα τη άμυνα και να ενισχυθεί η αμυντική βιομηχανία ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελέσει ισχυρότερο εταίρο στον στρατιωτικό τομέα και μάλιστα τα επόμενα δύο χρόνια προβλέπεται να δοθούν 500 εκατομμύρια μονάχα από την Κομισιό ενώ το υπόλοιπο 80% του συνολικού κόστου εν καιρό κρίση οικονομική θα καλεστούν να το πληρώσουν τα κράτη-μέλη. Εδώ ήθελα να θέσω και ένα θέμα ε, νομι, νομι, νομι, νομικό. Πρέπει να τονίσουμε πως το άρθρο 41, παράγραφος 2 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει ξεκάθαρα πως οι δαπάνε που προκύπτουν από επιχειρήσει που έχουν στρατιωτικέ ή αμυντικέ συνέπειε δεν πρέπει να χρεώνονται στον προπολογισμό τη Ένωση. Και όμω δυστυχώ αυτό που επιχειρείται σήμερα είναι με τη δικαιολογία του άρθρου 173 για τη βιομηχανική πολιτική. Εμεί αφιζητούμε την, λοιπόν την νομική βάση και αναμένουμε από την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου και από την Επιτροπή Νομικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να πράξουν το ίδιο. Ε, η ΓΚΟΕ NGL ζητά να αξιοποιηθεί το μεγάλο αυτό κονδύλι των 500 εκατομμυρίων για την πρόθεση της επαναβιομηχανοποίησης ιδιαίτερα στα κράτη που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση και τι νεοφιλεύθερε πολιτικέ λιτότητα. Ε, με τροπολογία που έχουμε καταθέσει, απορρίπτουμε την πρόταση που κατατέθηκε για στρατικοποίηση τη Ένωση και ζητάμε να κατατεθεί άμεσα πρόταση για ανάπτυξη μια ολοκληρωμένη βιομηχανική στρατηγική, η οποία να αντιμετωπίσει την ενεργεία, και να συμβάλλει στη βιώσιμη κοινωνική ανάπτυξη και στην ενίσχυση τη ποιότητα ζωή των λαών. Ιδιαίτερα προβληματισμό στην παρούσα πρόταση θεωρούμε το γεγονό ότι τα 500 εκατομμύρια που θα διατηρηθούν θα αποκοπούν από άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, προκαλώντα έτσι διπλή ζήμη. Για παράδειγμα, ενώ γίνεται συζήτηση για την ανάγκη ενίσχυση των προσπαθειών για ε, άσκηση τη απομόνωση των κρατών και περιοχών από τα ενεργειακά δίκτυα, για ενίσχυση ε, του προγράμματο συνδέοντα την Ευρώπη, εδώ προτείνονται να αποκομπούν 145 εκατομμύρια από αυτό το πρόγραμμα για να επιδηθούν στην αμυντική βιομηχανία και εμεί αυτό το θεωρούμε απαράδεκτο. Ε, στην τελική αυτό προτείνεται να αποκοπούν λεφτά από αναπτυξιακέ πολιτικές για να επενδυθούν στην ενίσχυση των αμυντικών και στρατηγικών δομών τη Ένωση. Γι' αυτό και η θέση μα είναι μια συνολική απόρριψη τη πρόταση όπως, ζητούμε ορισμένες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 is absolutely possible to speak in Greek. So um, you are replacing uh, Mr. Silikiotis and the floor is yours. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε τη δυνατότητα να διαβείς όπως είναι η τροποποίηση της οδηγίας για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου. Το ελάχιστο που επιβάλλει είναι να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για ολοκληρωμένη ανάλυση και ζωή παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να εκπονεί μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων για όλα τα νομοθετικά μέτρα που προτείνει, στην προκειμένη περίπτωση για εμάς είναι ξεκάθαρο πως η νέα οδηγία αποσκοπεί στην χειραγώγηση των κρατών μελών σχετικά με την ανάπτυξη αγωγών με τρίτες χώρες. Γι' αυτό λέμε ξεκάθαρα, αλλά και από το διεθνές δίκαιο. Έπειτα δεν γίνεται να μην λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες που υπάρχουν σε κάθε κράτος, οι οποίες καθιστούν αναντικατάστατο το ρόλο. Το μόνο που θα επιτύχει η νέα οδηγία είναι να αυξηθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ένωση στην ενεργειακή τροφοδοσία και ασφάλεια. Στα σοβαρά ενεργειακά προβλήματα και αδί... ώστε να τεθεί ο φραγμός στο Nord Stream 2. Οι τροπολογίες που θα καταθέσει η ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτική Αριστεράς θα αποσκοπούν στη διόρθωση